εσείς μια εισαγωγή, κάτι να τους πείτε να βγάλουν. Και ότι έχουμε την interpretation στις γλώσσες αυτές. So your attention please. Welcome to the European Parliament. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο σεμινάριο για τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με πολύ μεγάλη χαρά υποδέχομαι εδώ εσάς, τους δημοσιογράφους από τα κράτη-μέλη και ελπίζω ότι θα σας φανούν χρήσιμες οι συζητήσεις που θα ακολουθήσουν. Ελπίζω ότι θα γίνει επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων με την υπεύθυνη για τα θέματα επικοινωνίας, επικοινωνιακής πολιτικής αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου μας, την κυρία Κράτσα και του λοιπά μέλη ε, που θα είναι εδώ παρόντα. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως υπάρχει η διερμηνία στην αγγλική, γαλλική, ισπανική, ιταλική και ελληνική γλώσσα. Θα παρακαλέσω λοιπόν τώρα την κυρία Κράτσα, την αντιπρόεδρό μας, να κάνει την παρουσίαση, την εισήγηση. Καλημέρα σας, θα μιλήσω στα ελληνικά. Κυρίες και κύριοι, ε, με χαρά υποδεχόμαστε σήμερα τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης με, στο σεμινάριό μας με θέμα «Οι επιπτώσεις της συνθήκης της Λισαβόνας στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». Και επιτρέψτε μου, ως Ελληνίδα Ευρωβουλευτής, να κάνω και ειδική μνήμα στην παρουσία δημοσιογράφων προερχομένων από διάφορες περιοχές της χώρας μου και ιδιαίτερα από την ιδιαίτερα μου πατρίδα τη Ζάκυνθο. Κυρίες και κύριοι, το σεμινάριο αυτό αποτελεί μια από τις πρωτοβουλίες της Διεύθυνσης Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κ προείσταται της διεύθυνσης αυτής. Ε, ο στόχος της διεύθυνσης είναι η ενημέρωση των δημοσιογράφων επί θεμάτων της κοινοβουλευτικής μας δραστηριότητας αλλά και της ευρωπαϊκής επικαιρότητα γενικότερα. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω θερμά τους διοργανωτές που μας δίνουν την ευκαιρία της σημερινής εκδήλωσης. Κυρίες και κύριοι, μεταξύ των στόχων που έχω θέσει με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Αντιπροέδρου αρμόδιας για θέματα επικοινωνίας, κεντρική θέση έχει η ενημέρωση των δημοσιογράφων. Πιστεύω απόλυτα στη σημασία του ρόλου σας ως κοινωνών του μηνύματός μας στην κοινή γνώμη των κρατών μελών, όπως και σε ειδικέ κοινωνικο-επαγγελματικές ομάδες που δρούν σε επίπεδο εθνικό ή ευρωπαϊκό. Πιστεύω σε μια ανεξάρτητη δημοσιογραφία, αποτελεί αρχή της δημοκρατίας μας εξάλλου, μια δημοσιογραφία όμως που έχει τις δυνατότητες για να παρακολουθεί τις δραστηριότητές μας με κριτικό και δημιουργικό τρόπο. Παράλληλα θέλω να σας υπενθυμίσω ότι το ρόλο των δημοσιογράφων τον τιμάμε πολύπλευρα. Έχουμε θεσπίσει το βραβείο δημοσιογραφίας που απονέμουμε ετησίως για το σύνολο του ευρωπαϊκού τύπου, γραπτό, τηλεόραση, ράδιο, ίντερνετ και το οποίο παρουσιάζει όλο και περισσότερο ενδιαφέρον και συμμετοχή. Οι αρχές αυτές της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας αποτυπώνονται και σε άλλες μας δραστηριότητες. Παραδείγματος χάρη το βραβείο Ζαχάροφ που έχει θεσμοθετήσει εδώ και 20 χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να τιμήσει τους ανθρώπους που αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα πολλές φορές έχει απονεμηθεί σε δημοσιογράφους που με αντίξωες συνθήκες σε διάφορες περιοχές του κόσμου στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο αλλά και εκτός Ευρωπαϊκής Ήπειρου προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά του δημοσιογράφου. Ε, όπως γνωρίζετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες και ένα όλο και πιο εξειδικευμένο πρόγραμμα υπηρεσιών για να ε, κάνει αποτελεσματικές τις σχέσεις μας, τις σχέσεις του θεσμικού οργάνου, τις σχέσεις των ευρωβουλευτών με τους δημοσιογράφους, με τα μέσα ενημέρωση ευρύτερα έχει οθετήσει εδώ και χρόνια ένα πρόγραμμα προσκλήσεων εκπροσώπων του τύπου στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο προκειμένου να τους δώσει την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις εργασίες της Ολομέλειάς μας ή τις εργασίες κοινοβουλευτικών επιτροπών. Έχει οθετήσει επίσης πρόγραμμα σεμιναρίων στις περιφέρειες των χωρών μελών της Ένωσης, όπως και στις Βρυξέλλες, ε, γενικά για να διατηρήσει αυτή την ανταλλαγή απόψεων και να δώσει την ευκαιρία στα περιφερειακά μέσα να βρεθούν στο κέντρο της συζήτησης για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και το διακριτό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, στο πλαίσιο της λειτουργίας των κοινωνικών οργάνων λόγω του περιορισμένου χρόνου δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε περισσότερα παραδείγματα ε, και παρουσίαση των υπηρεσιών μας, διότι θα έχετε την ευκαιρία στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου αυτού να το παρακολουθήσετε από τους ε, αρμόδιους εκπροσώπους της Διεύθυνσης Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, θα ήθελα πάντως να σας πω ότι ε, τα μέσα που διαθέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, τα οπτικοακουστικά μέσα ε, τίθενται στη διάθεση των δημοσιογράφων για τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές εκπομπές και έχουν την δυνατότητα βέβαια σήμερα να παρακολουθήσουν τις εργασίες της Ελομέλειας και των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών μέσω δορυφόρου και υπολογιστή καθώς και μέσω του τηλεοπτικού μας ε, καναλιού. Και Ιδιαίτερα θέλω να αναφερθώ στην χρήση των μέσων επικοινωνίας μέσω διαδικτύου. Όλες αυτές οι πληροφορίες που θα έχετε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της συζήτησης του σεμιναρίου αυτού είναι πολύ χρήσιμες διότι όταν τις γνωρίζετε θα μπορέσετε να τις αξιοποιήσετε και για μας είναι πολύ μεγάλη, έχει μεγάλη σημασία να μπορέσετε να τις αξιοποιήσετε διότι μόνο τότε θα φέρετε την Ευρώπη και τη δημοκρατία πιο κοντά στους πολίτες. Κυρίε και κύριοι, η επικαιρότητα η ευρωπαϊκή σηματοδοτείται από την ε, θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία συμπίπτει παράλληλα με την 20η επέτειο από την πτώση του τείχους του Βερολίνου, κάτι που σηματοδότησε τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, αλλά και την ανάγκη για μια νέα διακυβέρνηση της Ένωσης όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κ. Μπούζεκ, η νέα συνθήκη προσφέρει λοιπόν για πρώτη φορά στην ιστορία της Ένωσης ένα πλέγμα δημοκρατικών και αποτελεσματικών κανόνων και διαδικασιών που δίνουν απαντήσεις στα προβλήματα 500 εκατομμυρίων πολιτών της Ένωσης. Αισθάνομαι ότι το ερώτημα που έχουμε να απαντήσουμε κι εσείς και εμείς είναι κοινό και συγκεκριμένο. Γιατί αυτή η νέα συνθήκη κάνει την Ένωση, όπως διαλαλούμε παντού, πιο δημοκρατική, πιο αποτελεσματική, πιο πολιτική. Η απάντηση είναι σαφής. βασικός λόγος είναι διότι παραχωρεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το μόνο άμεσα εκλεγμένο θεσμικό όργανο της Ένωσης μια σειρά νέων αποφασιστικών αρμοδιοτήτων αρμοδιοτήτων που εξασφαλίζουν ισοτιμία με το Συμβούλιο Υπουργών σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή νομοθετική διαδικασία. Σχεδόν το σύνολο του νομοθετικού έργου της Ένωσης θα αποφασίζεται από την 1η Δεκεμβρίου με βάση τη διαδικασία της συναπόφασης, διαδικασίας που διασφαλίζει ότι σχεδόν τίποτα πλέον δεν θα αποφασίζεται χωρίς την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 40 τομείς της κοινοτικής πολιτικής, επ' των το Κοινοβούλιο δεν είχε αποφασιστικό ρόλο, θα υπάγονται πια στην διαδικασία συναπόφασης. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας αναφέρω ορισμένα παραδείγματα επιμέρους πολιτικών που καθιστούν σαφή την αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τη νέα συνθήκη. Μια αρμοδιότητα κλειδί είναι αρμοδιότητα για την κοινή αγροτική πολιτική, η οποία μέχρι τώρα αποφασιζόταν, αποφασιζόταν από το Συμβούλιο Υπουργών. Για πρώτη φορά, τα μέλη του Κοινοβουλίου μπορούν να αποφασίζουν για τις ευρωπαϊκές αγροτικές πολιτικές και τις χρηματοδοτήσεις τους που καλύπτουν το 40 και παραπάνω της 100 του κοινοτικού προϋπολογισμού. Το σύνολο πλέον και όχι ένα μέρος του κοινοτικού προϋπολογισμού θα υιοθετείται και από τα δύο όργανα, και από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο Υπουργών. Άλλες ε, σημαντικές πολιτικές, όπως η μετανάστευση, η ασφάλεια ε, της παροχής ενέργειας, δικαστικές και εσωτερικές υποθέσεις, υγεία, τα διαφορετικά ταμεία, θα υπάγονται και αυτά στη διαδικασία συναπόφασης. Το Κοινοβούλιο αποκτά επίσης σημαντικές αρμοδιότητες στον τομέα της εξωτερικής, εξωτερικής πολιτικής ένωσης, διότι όλες οι διεθνείς συμφωνίες που θα συνάπτει η Ένωση, όπως οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, θα απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου. Και γνωρίζετε πόσο το Κοινοβούλιο θέτει τα θέματα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναπόσπαστο κομμάτι των εμπορικών συμφωνιών. Αποτελεί λοιπόν μια εγγύηση για την δημοκρατία και την ειρήνη στον κόσμο και την αποτύπωση των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ότι θα έχει να δώσει το δικό του αποφασιστικό ε, ε, λόγο έγκρισης για τη σύναψη τέτοιων συμφωνιών. Τέλος, το κοινοβούλιο μας αναβαθμίζεται και σε σχέση με τα άλλα ευρωπαϊκά όργανα αφού η επιλογή του προέδρου της ευρωπαϊκής επιτροπής θα πρέπει να γίνεται από το κοινοβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία και όχι απλή πλειοψηφία όπως συμβαίνει σήμερα και ο ύπατος εκπρόσωπος για τις εξωτερικές σχέσεις θα εγκρίνεται από το κοινοβούλιο όπως και οι άλλοι ε, επίτροποι. Δεν έχω την πρόθεση να σας αναφέρω άλλα παραδείγματα, ήθελα απλά το στίγμα της προσοχής να, να, τονίσω, διότι οι συνάδελφοι θα αναφερθούν σε αυτά στη συνέχεια, συνάδελφοι οι οποίοι συμμετέχουν αποφασιστικά στη διαδικασία υιοθέτηση της νέας συνθήκης, διαχρονικά έχουν παίξει ρόλο, όπως ο κύριος Jean-Luc ο οποίος δεν είναι μαζί μας, ο πρώην Πρωθυπουργός του Βελγίου, θα έρθει σε λίγο, ο κύριος Ντιούφ, ο συνάδελφος, ο κύριος Χογκερέη και θα έχετε επίση την ευκαιρία να ακούσετε και τον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Πιτέλα, ο οποίος μαζί με μένα προσωπικά και ένα αντιπρόεδρο άλλων, τον κύριο Βιντάλ Κουάντρας, είναι αρμόδιος για την συναπόφαση, την αρμόδιος για το ρόλο συναπόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το Συμβούλιο Υπουργών. Θα ήθελα να σας επισημάνω, κυρίες και κύριοι, ότι το Κοινοβούλιο έχει ε, ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία του για αυτή τη νέα πραγματικότητα που θα αναβαθμίσει το ρόλο του. Ενισχύει με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και πόρους τις σχετικές υπηρεσίες του. Προσαρμόζει τις δομές και τον τρόπο λειτουργίας του. Το πιο σημαντικό όμως είναι η πολιτική οριμότητα που πρέπει να επιδείξει ανταποκρινόμενο από τη μια μεριά στις επιδιώξεις των πολιτών που είναι συνεχώς αυξανόμενες για το ρόλο που μπορεί να παίξει το Ευρωπαϊκό mm. Κοινοβούλιο και από την άλλη μεριά στη θεσμική ισορροπία της Ένωσης, σε μια ισορροπία δηλαδή που θα πρέπει να παίξει το αναβαθμισμένο κοινοβούλιο με το διευρυμένο ρόλο μαζί με τα άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μέχρι σήμερα ιστορία του απέδειξε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέκεται στο ύψος των περιστάσεων αυτού του συνεχώς εξελισσόμενου και αναβαθμιζόμενου ρόλου του και ότι η πορεία του οφείλεται στη δική του φιλοδοξία, στη δική του διεκδίκηση με επιτυχία της συνεχούς αναβάθμισης και στη δική του καλή χρήση αυτής της συνεχώς διευρυνόμενης αρμοδιότητας που έχει. Καταλήγοντας, θέλω να εκφράσω την πεποίθηση ότι ένα κοινοβούλιο πιο δυνατό, με βαρύτερο και αποφασιστικότερο ρόλο, θα ελκύσει τους Ευρωπαίους πολίτες. Θα τους φέρει πιο κοντά στην πολιτική ευρωπαϊκή διαδικασία και θα συμβάλλει σε μια Ευρώπη πιο συμμετοχική. Έχουμε όμως ανάγκη και εσείς να προβάλλετε, εσείς οι εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης, αυτή την αλλαγή στην ισορροπία δυνάμεων, στην αλλαγή υπέρ του κοινοβουλευτισμού και υπέρ της δημοκρατίας. Και όσο περισσότερο προβάλλετε τον αναβαθμισμένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εσείς ξέρετε καλά ότι οι πολίτες, η κοινή γνώμη θα στέκονται με ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά που γράφετε και σε αυτά που εμείς κάνουμε και τη σημασία που έχουν για μια καλύτερη Ευρώπη. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Η αφρόα συμμετοχή σας δείχνει το ενδιαφέρον που έχετε για αυτή την ανταλλαγή απόψεων και την ενημέρωση και σας εύχομαι να έχετε μια ευχάριστη διαμονή και χρήσιμη στις Βρυξέλλες. Τώρα θα δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Τζάνι Πιτέλα και ευχαριστώ άλλη μια φορά τους συναδέλφους και τους υπηρεσίες του Κοινοβουλίου που είναι παρόντες και συμμετέχουν σε αυτό το σεμινάριο. Σας ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Κύριε Πιτέλα, έχετε το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο, την κυρία Κράτσα, για αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία και για την πλήρη και πολύ εύστοχη παρουσίασή της. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και να χαιρετήσω όλους εσάς και τους ε, Πριν από λίγη ώρα, ένας από τους συνεισηγητές μας, ο κύριος Άντρου Νταφ, απέστειλε ένα μήνυμα μέσω του οποίου είπε ουσιαστικά «Αντίο Νίκαια, καλωσόρισες Λισαβόνα». Πρόκειται για ένα μήνυμα πάρα πολύ όμορφο και συμπαθέ στον τρόπο που εκφράστηκε και γεμάτο ενθουσιασμό φυσικά. Και εγώ συμμερίζομαι αυτόν τον ενθουσιασμό, διότι εμείς έχουμε στην πλάτη μας 8 χρόνια μιας κατάστασης λίμπο. 8 χρόνια προσπαθεί η Ευρώπη να αποκτήσει νέους κανόνες, να έχει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο και νέα δυνατότητα λήψης αποφάσεων για τις μεγάλες προκλήσεις τις οποίες καλείται να, να απαντήσει σε έναν ολαιόνα αυξανόμενο κόσμο. Για 8 χρόνια λοιπόν βρισκόμασταν σε μια κατάσταση λίμπο, ζούσαμε με ψωμί και νερό και παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση παρά τη στέρηση δεν πέθανε, κατάφερε να αποκτήσει μια συνθήκη η οποία φυσικά δεν είναι το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, το οποίο εμείς ελπίζαμε, αλλά δεν πάβει να είναι ένα μέσο το οποίο περιλαμβάνει μία σειρά από μεγάλες καινοτομίε, όπως πολύ σωστά σας είπε η συνάδελφος κυρία Κράτσα, και εγώ δεν θα ήθελα εδώ να επαναλάβω τα όσα είπε για τις νέες εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τα νέα πρόσωπα του υπάτου εκπροσώπου για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, ε, τη νομική υπόσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, τη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τις νέες αρμοδιότητες που έχει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να σταθώ μόνο σε ένα σημείο. Το θέμα των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίου. Πρόκειται για ένα νευραλγικό σημείο, διότι Καταρχάς είχε εκλειφθεί ως αποδυνάμωση των λειτουργιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά εάν κάποιος διαβάσει το θέμα πιο επιστομή, επισταμένα θα διαπιστώσετε ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο θα ενισχύσει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και θα ενισχύσει και τη διαθεσμική συνεργασία. Από αύριο λοιπόν οποιαδήποτε απόφαση η οποία σχετίζεται με μια ευρωπαϊκή οδηγία θα αποσταέλεται προληπτικά στα εθνικά κοινοβούλια τα οποία θα έχουν 8 εβδομάδες στη διάθεσή τους προκειμένου να εκφράσουν την άποψή τους για το κατά πόσο γίνεται σεβαστή η αρχή της επικουρικότητας και η αρχή της αναλογικότητας. Πρόκειται για ένα τρόπο, κατά την άποψή μου, αποτελεσματικό, προκειμένου να είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη η συνεργασία μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μέχρι τούδε, οι ευρωπαϊκές οδηγίες μεταφέρονταν στην Εθνική Νομοθεσία. Και επομένως, η συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων ουσιαστικά αφορούσε μόνο την ε, κατιούσα φάση και όχι την ανιούσα φάση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Από εδώ και στο εξή δεν θα είναι πλέον έτσι τα πράγματα. Τα εθνικά κοινοβούλια θα καλούνται να συμμετάσχουν ακόμα και στην προπαρασκευαστική διαδικασία, στην ανιούσα φάση που σας ανέφερα. Επομένω, η απόσταση μεταξύ πολιτών και θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μειωθεί αναγκαστικά. Αυτό θα είναι ένα σημείο το οποίο θα προσεγγίσει ακόμα περισσότερο τους Ευρωπαίου πολίτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από σήμερα το 70 με 75% της εθνικής νομοθεσίας καθορίζεται και επηρεάζεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και αυτό φυσικά θα αυξηθεί στο μέλλον και κυρίως θα είναι μια αμφίδρομη διαδικασία, αμοιβαία διαδικασία, η οποία σαφώς θα ωφελήσει και την ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και την εθνική νομοθεσία. Αυτό για μας σημαίνει ότι θα υπάρχει ε, μία νέα ευθύνη, μία ε, κατηγορηματική ανάγκη να κάνουμε πολύ καλύτερα τη δουλειά μας ως Ευρωπαίοι νομοθέτες, ε, αλλά σημαίνει επίσης και για μια, μια κατηγορηματική ανάγκη για όλους εσάς, για τους πολίτες, για τους πολιτικούς, για τους οικονομικούς φορείς και για τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι οποίοι δεν θα μπορούν πλέον να βλέπουν την Ευρώπη μόνο ως μια απομακρυσμένη πραγματικότητα ή μια πραγματικότητα στην οποία ορισμένες φορές έρχεται ένας τυχαίος να μας περιγράψει με στον φόδες ύφος και με διάφορα χρώματα ε, την Ευρώπη. Η Ευρώπη ελπίζω και πιστεύω θα είναι όλο ένα και περισσότερο αντικείμενο της προσοχής σας. Δεν σας ζητούμε μια προσοχή φιλική, συμβατική. Σας ζητάμε να μας κοιτάξετε με επικριτικό βλέμμα. Θέλουμε να μας παρακολουθήσετε, να μας εποπτεύετε και θέλουμε στις εφημερίδες σας και στις τηλεοράσεις σας τα ευρωπαϊκά θέματα να μην είναι θέματα εξωτερικής πολιτικής, διότι η Ευρώπη, η ευρωπαϊκή πολιτική είναι εσωτερική πολιτική για κάθε μία από τις χώρες μας. Επομένως, θα πρέπει να είναι εσωτερική πολιτική για όλα τα εθνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντιπρόεδρε. Και τώρα το λόγο θα δώσω στον Άρτη Αφιχθέντα, τον κύριο Λουκ Ντεάν, εκλεκτό συνάδελφο και πρώην Πρωθυπουργό του Βελγίου που έχει ασχοληθεί, όπως σας είπα στην αρχή, με την ε, θέση του Κοινοβουλίου για την ε, υιοθέτηση της συνθήκης Λισαβόνας και την εφαρμογή του στην ε, λειτουργία μας. Έχετε το λόγο, κυρία Πρωθυπουργέ. Uh, good afternoon. Uh, Καλησπέρα σας. Η συνθήκη της Λισαβόνας που θα τεθεί σε ισχύ από αύριο είναι, πιστεύω, ένα πολύ σημαντικό βήμα προόδου για την Ευρωπαϊκή Ένωση. είναι από αυτές τις συνθήκες που αποτελούν άλμα, θα έλεγα, μεγάλο άλμα, όπως η συνθήκη της Ρώμης, όπως το Μάστριχτ, όπως και η Λισαβόνα. Θα μας βοηθήσει λοιπόν να οργανώσουμε την Ευρώπη κατά τρόπο αποτελεσματικό και δημοκρατικό. Μια Ευρώπη με 25 κράτη-μέλη, μια Ευρώπη που θα είναι πραγματικά, πραγματικός ε, παράγουν στη διεθνή σκηνή ταυτόχρονα. Καθιστά λοιπόν την Ευρώπη και πιο δημοκρατική και πιο αποτελεσματική. Και εδώ ιδιαίτερη σημασία έχει να υπογραμμίσουμε την βασική αρχή που εγγράφεται στη συνθήκη πως η λήψη αποφάσεων στην Ευρώπη πλέον ακολουθεί τη μέθοδο της πλειοψηφίας πλην της έγκρισης συνθήκων. Ε, υπάρχουν φυσικά εξαιρέσεις στον βασικό κανόνα της πλειοψηφικής λήψης αποφάσεων, αλλά η ουσία είναι ότι υπάρχει αυτός ο κανόνας. Η παράδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπαγορεύει πλειοψηφικές αποφάσει να λαμβάνονται σε διαδικασία συναπόφαση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εφόσον λοιπόν υπάρχει πλειοψηφία, αναπτύσσεται διαδικασία συναπόφαση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι συμμετέχουμε και εμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με ιδιαίτερη σημασία στο γεγονό ότι αυτή η διαδικασία, αυτή η μέθοδο εφαρμόζεται και για τον προπολογισμό, πράγμα που δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Υπάρχει επίση ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο θα έλεγα βρίσκεται μεταξύ των ενιών του, της αποτελεσματικότερης μεθόδου εργασίας και της παρουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην, Ευρω... στη διεθνή σκηνή, είναι ότι διευκρινίζονται πλέον οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πέραν αυτού προστίθενται στο κατάλογο αρμοδιοτήτων της και νέες. Θα ήθελα λοιπόν να σας αναφέρω μερικές από αυτές. Η ενέργεια καταρχάς. Αποκλειστική πλέον, γιατί μέχρι τώρα ήταν συντρέχουσα αρμοδιότητα, Μέχρι τώρα δηλαδή η Ευρώπη συνέδεε την ενέργεια με το περιβάλλον ή με τις αγορές, με τα θέματα της ελεύθερης αγοράς, αλλά δεν ήταν αποκλειστική αρμοδιότητα. Το ίδιο ισχύει και για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Σημαντικό βήμα επίσης αποτελεί το γεγονός ότι ο τρίτος πυλώνας, δικαιοσύνη και εσωτερικά, κατά κανόνα πλέον, υπάγεται επίσης στις κοινοτικέ αρμοδιότητες. Αποτελεί ύλη νομοθετική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με πάλι πολύ σημαντικό ρόλο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο πλέον αναλαμβάνει ως Ευρωπαίος νομοθέτης δράση, γιατί οι αποφάσεις πλέον λαμβάνονται στο ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι σε διακυβερνητικό επίπεδο μεταξύ κυβερνήσεων. Άλλο ένα πολύ σημαντικό στοιχείο λοιπόν ενίσχυσης του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τρίτο στοιχείο. Η Ευρώπη ως παράγον στη διεθνή σκηνή. Εδώ νομίζω συμφωνούν όλοι πως η Ευρώπη είναι ισχυρότερη όταν μιλάει με μία φωνή ενωμένη. Το πρόβλημα όμως είναι ότι η Ευρώπη, εάν δεν έχει προβλεφθεί στην οργάνωσή της, δεν μιλάει συνήθως με μία φωνή. Δεν εκφράζεται ενωμένα. Ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτού είναι ο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου ασφαλώ. Θα πρέπει πιστεύω όμως να επιδιώξουμε με τον ίδιο ε, νοτικό τρόπο να δρούμε σε άλλα διεθνή φόρα, σε άλλους διεθνείς φορείς και οργανισμούς. Και πάλι εδώ χρειάζεται οργάνωση, δεν γίνεται δηλαδή αυθόρμητα αυτή η μετάβαση και δεν είναι και εύκολη. Φερρυπίν, υπάρχουν πολλές δυνατότητες που προβλέπονται μέσα από τη συνθήκη ώστε η νομισματική ένωση να δρά ως ένωση, να δρά δηλαδή ως μία φωνή μέσα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όμως αυτό δεν συμβαίνει. Δεν έχουμε καταφέρει να το κάνουμε αυτό. Χρειάζεται λοιπόν μια εσωτερική δυναμική να αναπτυχθεί που θα μας επιτρέψει και προς τα έξω να ε, μιλάμε ως ένα πρόσωπο, ως ένας φορέας, ως ένας παράγων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί και κατά την συντακτική ε, διάσκεψη κατέστη πολύ σαφές ότι θα παραμείνουν οι εξωτερικές δράσεις αντικείμενο ε, διακυβερνητικής συνεργασίας, όμως επιδιώκαμε από την αρχή να μην είναι αντικρουόμενες οι εξωτερικές πολιτικές. Δηλαδή η Επιτροπή και το Συμβούλιο να ακολουθούν την ίδια γραμμή. Έτσι λοιπόν η δικέφαλη αρχή με τον είπα το εκπρόσωπο για τα εξωτερικά και τον πρόεδρο ε, έχει πολύ μεγάλη σημασία αφενός με την έννοια της συνέχειας ο Χαβιέρης Σενσολάνο, ο οποίος δεν ήταν υπέρ της δικέφαλης αρχής αλλά επεδίωκε να αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου Εξωτερικών, τώρα λέει, ε, μάλλον έλεγε ως επιχείρημα ότι κάθε φορά που ξεκινάει μια εξάμηνη εναλλασσόμενη Προεδρία πρέπει να ξεκινήσουμε ε, και την επεξεργασία του προγράμματος του επόμενου εξαμήνου. Γιατί δεν μπορούμε βέβαια να γελιοποιούμαστε στη Ουάσιγκτον και εδώ και εκεί όπου έχουμε να πάμε. Πράγμα το οποίο έλεγε ο Σολάνο, εμένα δεν με βοηθάει καθόλου στη δουλειά μου γιατί δεν μπορώ να παρακολουθήσω τα τρέχοντα θέματα έχοντα υπόψη μου τι θα γίνει μετά. Τώρα λοιπόν και δεδομένου ότι τα μέσα, τα πρακτικά, οι δυνατότητε είναι στα χέρια τη Κομισιόν, πρέπει να έχουμε αυτή τη δυνατότητα στο επίπεδο τη Κομισιόν. Αυτό γίνεται τώρα, δηλαδή η εξωτερική υπηρεσία αυτή, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση κοινή για το Συμβούλιο και την Κομισιόν εδρεύει στην Κομισιόν. Με αυτήν αναπτύσσεται μια ευρωπαϊκή πολιτική που μέχρι στιγμής μόνο είναι πολιτική αντιμετώπισης κρίσεων. και ασφαλώς με την ανάπτυξη των αντιπροσωπιών και των πρεσβειών στο, στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου μπορούμε να έχουμε πιο καλή παρουσία και αποτελεσματικότητα. Ταυτόχρονα δε και το Κοινοβούλιο μπορεί, όχι άμεσα βέβαια για την εξωτερική πολιτική, γιατί όπω είπα παραμένει σε επίπεδο διακυβερνητική συνεργασία, διακυβερνητική πολιτική, έμεσα στον προπολογισμό, δηλαδή εκεί που προσδιορίζονται οι πόροι που διατίθενται ή απελευθερώνονται για χρήση σε ε, θέματα εξωτερικής πολιτικής. Το Κοινοβούλιο λοιπόν μπορεί επειδή απαιτείται η δική του έγκριση για να αποδεσμευθούν τα κονδύλια, να έχει ένα λόγο και στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Οι τρεις στόχοι λοιπόν που επιδιώξαμε με τη συνθήκη, η αποτελεσματικότητα με 27 κράτη-μέλη, πιο δημοκρατική οργάνωση και η πιο κοινοτική προσέγγιση με πιο πολλούς κοινού τομείς, αλλά και η οργάνωσή μας, η οργάνωση Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ενός διεθνούς παράγοντα, ενός παράγοντα στη διεθνή σκηνή που να μπορεί να μιλάει με μια φωνή. Αυτοί οι στόχοι λοιπόν έχουν, επιτυχθεί έχουν επιτευχθεί σε σημαντικό βαθμό από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Έχει επιτύχει δηλαδή η συνθήκη της Λισαβόνας μεγάλα βήματα στους τρεις αυτούς τομείς και ταυτόχρονα εξασφαλίζει και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο με τη διαδικασία της συναπόφασης με την κοινοτική μέθοδο και μέσω του προϋπολογισμού για τα εξωτερικά, για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε από πλευρά μα εντωμεταξύ αναλάβει μια τεράστια ευθύνη. Είναι μεγάλη η πρόκληση που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ε, υλοποιήσει, να οργανώσει καταρχά, να οργανωθεί το, στο εσωτερικό του, να οργανώσει ιστορικά τι υπηρεσίε του, γιατί χωρί αυτό δεν θα τα καταφέρει ποτέ βέβαια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντεάν. Ο λόγος τώρα στον κύριο Άντριο Ντάφ, ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων για εκ της Ομάδας των Φιλελευθέρων για την Ευρώπη και υπήρξε εισηγητέ ε, σε κάποια ουσιαστικά θέματα της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων για τη συνθήκη της Λισαβόνας και για την ε, περίοδο πριν από την ε, κύρωση της συνθήκης της Λισαβόνας. Παρακαλώ. Good afternoon, everyone. Um, Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Και πρόκειται για μια εξαίρετη ευκαιρία, πιστεύω, σήμερα να συστήσουμε τη νέα συνθήκη. Το Κοινοβούλιο, όπως και όλοι πιστεύω, περάσαμε πολύ καιρό ανησυχώντας, σκεπτόμενοι, αναλογιζόμενοι, προσπαθώντας να βρούμε μια λύση, μια νέα διαδικασία που θα μπορούσε να φέρει κοντά, να καταστήσει συνομιλητές και τους λαούς αλλά και τα 27 εθνικά κοινοβούλια. Λόγω αυτής της ε, αμφιβολίας, αβεβαιότητας που επικράτησε, ε, χάσαμε λίγο την ουσία. Δεν ασχοληθήκαμε δηλαδή με την ουσία και το επίτευγμα το βασικότερο αυτής της νέα συνθήκη, ότι δηλαδή εξασφαλίζει περισσότερη ολοκλήρωση ευρωπαϊκή. Και ιδιαίτερα συμφωνώ με την εκτίμηση του Ζων Λουκ Αν ότι πρόκειται για μια ιστορική συνθήκη, για ένα ιστορικό άλμα. Ένα άλμα το οποίο θα πρέπει βεβαίως και να εκτιμήσουμε στις σωστές του διαστάσεις, αλλά που δεν πρέπει να λησμονούμε ότι εμείς ως Κοινοβούλιο έχουμε περισσότερες πλέον εξουσίες και είναι στο χέρι μας εντό εισαγωγικών να κερδίσουμε περισσότερες, περισσότερο σεβασμό καθώς είμαστε πλέον πιο υπεύθυνοι μέσα από τη διαδικασία του προϋπολογισμού και τη ε, την ομοπαραγωγική διαδικασία. Δεν είναι υπερβολή νομίζω. Το να πούμε ότι βρισκόμαστε σε μια κοινοβουλευτική πλέον δημοκρατία. Μια ομόσπονδη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αυτό καταφέραμε να δημιουργήσουμε, να οικοδομήσουμε. Αυτό δεν το λέω μόνο και μόνο γιατί ενισχυθήκαν οι εξουσίες του Κοινοβουλίου. Όταν αναλογιστούμε το πώς άλλαξαν λειτουργία, ύφος, νοοτροπία ακόμη ε, τα μέλη του Συμβουλίου, η συμπεριφορά του Συμβουλίου πώς άλλαξε, νομίζω αντιλαμβάνεται κανείς ότι έχουμε μεγάλες αλλαγές, γιατί το Συμβούλιο πλέον εκτίθεται και στον έλεγχο του τύπου. Πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ δηλαδή ο τύπος να είναι σε θέση να παρακολουθήσει μέσα από το κτίριο, μέσα από τις αίθουσες του Συμβουλίου, τις συνεδριάσεις του. Θα δείτε ότι το Συμβούλιο θα υποχρεωθεί να μπει σε δεύτερη μοίρα, να συμπεριφερθεί ως μία άνοβουλη ως μια ένα δεύτερο δηλαδή νομοθετικό σώμα ενός κράτους ως μια γερουσία ενώ μέχρι τώρα συμπεριφερόταν περισσότερο μια διάσκεψη διπλωματική. Ο Τζάνι Πιτέλα μίλησε νωρίτερα για, την, για τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες των Εθνικών Κοινοβουλίων που επίσης θα πρέπει να σημειώσουμε ενισχύονται και θα πρέπει να αξιοποιηθούν στον ορθό βαθμό από τους ε, εθνικούς βουλευτές. Προσπαθήσαμε επίσης να προστεύσουμε ή με τι άλλο να διευκρινίσουμε τις πολιτικές διαδικασίες που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα πιστεύω πρέπει να εμφυσίσουμε πνεύμα πολιτικό, πνεύμα πολιτικής στο συνταγματικό οικοδόμημα, στην ε, συνταγματική μας δομή. Ένα κύριο ζήτημα που θα πρέπει να μελετηθεί προσεκτικά είναι η συνεργασία, καλύτερα ο συντονισμός μεταξύ των τεσσάρων προσώπων που μοιράζονται τις ύπατες εξουσίες, τα ύπατα αξιώματα της δομής αυτής. Γιατί βέβαια έχουμε ασφαλώς τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον πρόεδρο του Συμβουλίου, τον εκπρόσωπο για τα εξωτερικά, την εκπρόσωπο, την καθημερινά αλλά ως τέταρτο τον προ, ε, προεδρεύοντα, το Πρωθυπουργό δηλαδή της ε, Προεδρίας, ο οποίος έχει πολύ σημαντικό ρόλο συντονισμού του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων. Το οποίο αποκόπτεται από το Συμβούλιο των Εξωτερικών. Αυτό που προσπαθούμε να επιτύχουμε, βεβαίως, είναι να να εξασφαλίσουμε το ότι οι Υπουργοί των Εξωτερικών θα ασχολούνται με την εξωτερική πολιτική, όπως οφείλουν, και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε τον εσωτερικό συντονισμό του Συμβουλίου, ο οποίος ήταν μάλλον ελλειπής ή αδέξιος μέχρι τώρα. Αυτή, αυτά τα τέσσερα πρόσωπα λοιπόν, θα έλεγα το G4 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να ε, αναπτύξουν μεταξύ τους ένα ικανοποιητικό επίπεδο συνεννόησης και συνεργασίας, πράγμα το οποίο μέχρι στιγμής δεν είχαμε. Στο εγγύς μέλλον, ο κύριος τομέας που θα δούμε όπου θα δούμε πολύ γρήγορα εξελίξει που θα προσθέσει μεγαλύτερε μεταλλάξει, θα είναι το μέσο εξωτερική πολιτική και τη πολιτική ασφάλεια. Και εδώ νομίζω θα δούμε πολύ γρήγορα τα πρώτα μηνύματα που προετοιμάζουν μερικά κράτη και που θα εκδηλωθούν ως ένας πρώτος πυρήνας κρατών στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας για την δημιουργία μιας μόνιμης δομής, μιας πιο ολοκληρωμένης δομής στην άμυνα όπου φυσικά τίθεται το ερώτημα του τι στάση θα τηρήσει η Μεγάλη Βρετανία εάν θα επιλέξει να μείνει στο περιθώριο εάν προτιμήσει δηλαδή να μείνει εκτός αυτής της νέας εξέλιξης πράγμα το οποίο είναι δική της επιλογή αλλά όταν αναπτύσσετε ένας άξονας Βερολίνου-Παρισίων καθίσατε ασφαλώς αισθητή η απουσία του Λονδίνου το οποίο όμως ταυτόχρονα μένοντας έξω από το χορό δεν θα μπορεί και να παρεμποδίσει την δημιουργία ενός τέτοιου πυρήνα, μιας ομάδας κρατών που θα θέλουν να προχωρήσουν πιο γρήγορα στα θέματα αυτά της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας. Μια άλλη μεγάλη πολιτική πρόκληση για μας. Μια πρόκληση που δύσκολα πιστεύω θα φέρουμε εις πέρας. Είναι το ζήτημα των ε, δημοσιονομικών δομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε ότι έχουμε ενόψει μια δημοσιονομική μεταρρύθμιση, πρέπει να ολοκληρωθεί πριν το 2014, Φρονώ δε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, άκρος δυσχερές για τα 27 κράτη-μέλη, το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, βρούνε μια λύση. Μιλήσουμε μονούμε ότι ως παράγον αυτών των αποφάσεων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει και θα πρέπει να ε, συμβάλλει στην εξέβρεση συμφωνίας. Πολλέ φορές έχουμε δει σε περιπτώσεις όπου κάποια απόφαση δυσκολευόταν να εγκριθεί, ήταν δύσκολο να εγκριθεί, όπως με τις οδηγίες ε, για τις υπηρεσίες ή για τα χημικά, βλέπαμε ότι τα προβλήματα εντοπίζονταν περισσότερο σε επίπεδο συμβουλίου, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πολύ πιο πρόσφορος ε, συνομιλητής για την ε, εξέβρεση λύσης. Καθώς όμως τα προβλήματα τα οικονομικά επιδεινώνονται καθώς συρρυκνώνεται το ΑΕΠ μας και αντιμετωπίζουν οι πολίτες μας περισσότερα οικονομικά προβλήματα, θα υπάρχουν μάλλον δυσκολίες στην ενίσχυση του προϋπολογισμού και οι μεταφορές κονδυλίων από τα κράτη-μέλη στον κοινό προϋπολογισμό για κέριους τομείς δαπανών θα περιοριστούν ή θα πρέπει να είναι στοχευμένα περισσότερο στην έννοια του, ε, της ικανοποίησης με τον καλύτερο τρόπο ενός καλού αποτελέσματος. Δηλαδή θα γίνεται ο έλεγχος του ε, κόστους και του αποτελέσματος εκεί που δηλαδή η διάθεση των κονδυλίων εξασφαλίζει οικονομίες κλίμακος. Εδώ θα δοκιμαστεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως προς την αποτελεσματικότητά του, ως προς τον τρόπο λειτουργίας του. Πρόκειται για μια πρόκληση την οποία πιστεύω είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε και πιστεύω ότι η εμπιστοσύνη αλλά και η αυτοπεποίθησή μας θα ενισχυθούν. Η εμπιστοσύνη που έχουν για μας οι πολίτες, η δική μας αυτοπεποίθηση θα ενισχυθούν μετά την θέση σε ισχύ αυτής της νέας συνθήκης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και για να ολοκληρώσουμε αυτό τον πρώτο γύρο παρεμβάσεων να δώσω το λόγο στο Ρωμόν Χαουρεγγί, ο οποίος είναι ο συντονιστής των ε, Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Να ευχαριστήσω και την Αντιπρόεδρο για την ε, πρόσκληση. Θα ήθελα Καταρχάς, να μοιραστώ μαζί σας ένα παράδοξο. Τις τελευταίες εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε τέσσερις πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις. Όπως είπαμε εδώ, ίσως ιστορικές. Αύριο τίθεται σε ισχύ η νέα συνθήκη, ε, βάζοντας τέλος σε 8 χρόνια βεβαιότητας. Εκλέξαμε πρόεδρο της ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπής με πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μετά από ομόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχουμε πλέον μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία ανακοινώθηκε την περασμένη Παρασκευή και για πρώτη φορά επιπλέον το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέλεξε πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπα το εκπρόσωπο για τις εξωτερικές σχέσεις. Πρόκειται λοιπόν για τέσσερις πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις. Ωστόσο, διερωτούμε γιατί υπάρχει τέτοια απαγοήτευση στην Ευρώπη. Ένας γνωστός Βρετανός ακαδημαϊκός, ευρωπαϊστής, ε, σε ένα από τα άρθρα τα οποία πολύ συχνά δημοσιεύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έβαλε τίτλο «Πώς φτάσαμε σε αυτό». Έτσι έλεγε ο Γκόρντον Άσ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε τόσες μεγάλες προόδους σε τέσσερις λίγες εβδομάδες υπάρχει τόσο μεγάλη απεσιοδοξία για το μέλλον της Ευρώπης. Πιστεύω ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο μας αφορά όλους, κυρίως ε, αυτή τη στιγμή που συζητάμε, διότι νομίζω ότι ξεκινάει μια νέα πορεία για την Ευρώπη. Έχουμε μια νέα αρχιτεκτονική δομή, ένα νέο ε, νομικό ε, και πολιτικό μέσο. Έχουμε νέες αποφάσεις. Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω τρεις ε, σκέψεις μου για να τηρήσω και τα χρονικά περιφέρεια, τα οποία θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά θέματα από τούδε και στο εξής. Καταρχά, η συνθήκη τη Λισαβόνα είναι απαραίτητη συνθήκη προκειμένου να υπάρξει πρόοδο στην Ευρώπη, αλλά δεν είναι ικανή συνθήκη. Η συνθήκη τη Λισαβόνα δίνει τη δυνατότητα, δίνει τα μέσα για να μπορέσουμε να προοδεύσουμε στην ολοκλήρωση και στο να είμαστε Ευρωπαίοι αλλά λείπει η πολιτική βούληση. Το πνεύμα το οποίο έδωσε ε, ζωή στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν ήταν ακόμα στα Σπάργανα θα πρέπει ίσως να αναθεωρηθεί. Το πνεύμα της δημιουργίας ενός χώρου ο οποίος ε, θα βασίζεται στην ειρήνη βάσει της ιστορικής μνήμης του πολέμου ή των πολέμων ε, είναι ερώτημα τύπου Άμλετ. Να ζει κανεί ή να μη ζει. Όπω έλεγε ο Χαβιέρ Σολάνα σε μια συνέντευξη σήμερα, σημαίνει το να είναι κάποιο παγκόσμιο παίκτη. Διότι αν δεν είμαστε παγκόσμιοι παίκτε, δεν είμαστε στην Ευρώπη. Στη νέα διακυβέρνηση του κόσμου, ε, στι νέε θέσει τι οποίε είναι παρούσα η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή θα είναι η Ευρώπη ή δεν υπάρχουμε. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο ζήτημα το οποίο ε, δημιουργεί σκέψεις ως προς το ρόλο του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να μιλάμε με μια ενιαία φωνή, με αυτή τη νέα συνθήκη, σε αυτό το νέο χώρο τον οποίο ε, έχουμε αυτή τη στιγμή. Η δεύτερη σκέψη αφορά εμάς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι συνάδελφοι λογικά είπαν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλάζει εκ απορροφά ένα σύνολο νομοθετικών ε, λειτουργιών πλέον, αλλά αυτό θα πρέπει να δημιουργήσει και σκέψεις στις πολιτικές ομάδες, σε εμάς τους ίδιους. Διότι εκεί που ήμασταν μια βουλή που ετοίμαζε γνωμοδοτήσεις για να εισακουστούμε, γινόμαστε πλέον νομοθέτες. Έχουμε πλέον την αίσθηση ευθύνη που ε, έχει ο, αυτός ο οποίος κυβερνά. Και αυτό φυσικά θα αλλάξει ριζικά το ρόλο μας, τον τρόπο με τον οποίο ε, ετοιμάζουμε τις νομοθετικές μας πράξεις και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το σκεφτεί πολύ σοβαρά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να το προσφέρουμε και σε εσά, ε, διότι είμαστε πρώτον πυλών τη θέση σε ισχύ τη ε, συνθήκη τη Λισαβόνα. Όπω είπε πολύ σωστά ο Τζάνι Πιτέλα, θα πρέπει να σκεφτούμε επίση και το νέο ρόλο που θα έχουν τα εθνικά κοινοβούλια ως προσπιστές θεματοφύλακες της αρχή της επικουρικότητας. Διότι η συνθήκη της Λισαβόνα δημιουργεί μια διαδικασία μέσω τη οποίας τα εθνικά κοινοβούλια ίσως σε κάποιες χώρες ε, και τα περιφερειακά κοινοβούλια με νομοθετικές αρμοδιότητες, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στην Ισπανία ή στις ομοσπονδιακές χώρες ή και στην Ιταλία, θα πρέπει να μπορούν να παρέμβουν σε μια διαδικασία προάσπιστης της αρχής επικουρικότητας η οποία εμπνέεται από τη συνθήκη και η οποία εμπνέει και το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Σα ευχηθώ την προσοχή όμω εδώ. Η αρχή της επικουρικότητας θα πρέπει να εκλαμβάνεται με το σωστό τρόπο. Εάν ε, χρησιμοποιούμε κριτήρια φονταμενταλιστικά και προσεχή εδώ υπάρχουν πάρα πολλά ε, στοιχεία τέτοια, ε, θα οδηγηθούμε στην κατάρρευση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. θα πρέπει σε πάρα πολλές περιπτώσεις να αναγνωρίζουμε ότι πάβει να υπάρχει κυριαρχία. Εκχωρείται η κυριαρχία. Επομένω, και με αυτό θα ολοκληρώσω, πιστεύω ότι η εφαρμογή αυτού του νέου μηχανισμού παρέμβασης από πλευράς Εθνικών Κοινοβουλίων θα πρέπει να γίνεται με ευέλικτο τρόπο, ώστε να μην διαιωνίζονται οι διαδικασίες και να μην παραμένουν κενό γράμμα και με μέτρο. Διότι αν έχουμε ε, υπερβολή στην διατήρηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, δεν θα μπορεί ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προοδεύσει. Επί παραδείγματα, δείτε το χώρο ελευθερίας και δικαιοσύνης. Εδώ θα πρέπει να έχουμε ε, υπόψη ότι έχουμε πάρα πολύ διαφορετικά ποινικά συστήματα, διαδικαστικά συστήματα, αλλά για να προοδεύσουμε σε ένα χώρο ελευθερίας και δικαιοσύνης θα πρέπει να αρχίσουμε να ενοποιούμε κανόνες εάν ισχύει το κριτήριο της επικουρικότητας λαμβάνοντας υπόψη το, το, την κυριαρχία μας και μόνο δεν θα μπορέσουμε να προοδεύσουμε. Γι' αυτό εδώ θα πρέπει να σας ε, επιστήσω την προσοχή και να σας πω ότι θα πρέπει να γίνεται υπεύθυνα η χρήση της αρχής αυτής. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα νομίζω ότι έχουμε λίγο χρόνο στη θέση μα ακόμη για να υποβάλλετε τι ερωτήσει σα στου βουλευτέ. Ξέρω ότι κάποιοι από αυτού θα χρειαστεί να αποχωρήσουν ίσω λίγο νωρίτερα, αλλά θα προσπαθήσουμε να διαθέσουμε χρόνο για έρωτα ερωταποκρίσει, τουλάχιστον για 10-15 λεπτά και μετά να περάσουμε στο δεύτερο κομμάτι του σεμιναρίου. Παρακαλώ, κύριε Φρονκόλ. Σα παρακαλώ να μα λέτε πάντοτε το όνομά σα. και σε ποιον απευθύνεστε. Πέτερ Φων Κούλ από την Δανία. Θα ήθελα Καταρχάς, να σημειώσω ότι με έκπληξη διαπιστώνω ότι όχι μόνο αυξάνεται ο αριθμό των ε, βουλευτών, αλλά και του προσωπικού σας. Ποιος θα πληρώσει την ύφη, ο φορολογούμενος. Και δεύτερον, λέτε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να συνεργάζεται με τα Εθνικά Κοινοβούλια στα θέματα των εξωτερικών. Φερρυπίνε. Ε, το πρόβλημα με το Ιράν, το πρόβλημα το Παλαιστινιακό, σχέση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων, Αφγανιστάν, Τουρκία. Η, ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ζήτημα που θα κριθεί από το Κοινοβούλιο, από τον Πρόεδρο που έχει εκφραστεί δικατά, από τους Γάλλους που ζητούν δημοψήφισμα. Πώς εκφράζεται η μία φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιος ήθελε παρακαλώ να απαντήσει. <coughs> Uh, Ας ξεκινήσω εγώ και συνεχίζετε αν θέλετε για να δώσω απάντηση πρώτα στην τελευταία σας ερώτηση. Δεν αλλάζει τίποτα η συνθήκη ως προς την ένταξη νέων κρατών. Ακόμα η διαδικασία προβλέπει πως τη διαπραγμάτευση την κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έκθεση της την εγκρίνει το Συμβούλιο με τη μορφή μιας συνθήκης την οποία συνθήκη πρέπει να κυρώσει το κάθε κράτος μέλος με τις μεθόδους που προβλέπει το κάθε σύνταγμα. Με βάση τη σταγματική του τάξη. Παράδειγμα. Μιλήσατε για τη Γαλλία. Εάν η Γαλλία αποφασίσει ότι, αντίθετα με ό,τι έχει πράξει το παρελθόν, αυτή τη φορά θα χρειαστεί δημοψήφισμα, είναι δική της ευθύνη. Δεν θα παρέμβει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τρόπο ε, που θα ε, χρησιμοποιήσει το κάθε κράτο μέλο για την κύρωση της νέας συνθήκης, της, ε, της συνθήκης ένταξης. Και το Κοινοβούλιο επίσης έχει ρόλο να διαδραματίσει ως προς το ότι απαιτείται να γνωμοδοτήσει για τις συνθήκες ένταξης, αντίθετα από ό,τι συμβαίνει με την συνθήκη της το πρόβλημα στο οποίο αναφερθήκατε, αναγνώριση του, του κοσφοπεδίου και τα λοιπά διεθνή προβλήματα. Παραμένουν διακυβερνητικά, θέματα διακυβερνητικής συνεργασίας. Πλην όμως, με καλό συντονισμό της εξωτερικής πολιτικής, μπορούμε ενδεχομένως να βρούμε λύσεις στις οποίες να είναι σύμφωνα όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωση. Ωστόσο, το παρελθόν έχει αποδείξει ότι όπου είναι διακυβερνητική μέθοδος μπορούν κάποια κράτη-μέλη να προχωρήσουν χωρίς να περιμένουν τη συμφωνία των πάντων. Εγώ ελπίζω ότι η υπηρεσία εξωτερικών σχέσεων, ε, η δικέφαλη, προσώπηση περιπτώσει, ε, εκπροσώπηση της Ένωσης πλέον σε αυτό το επίπεδο, θα μπορέσει να πιέσει περισσότερο για από κοινού αντιμετώπιση των ζητημάτων. Αλλά ε, η συνθήκη δεν το επιβάλλει αυτό ως υποχρέωση και όπως είπα και νωρίτερα και πιστεύω ότι αυτό θα έχει κέρια σημασία στα επόμενα χρόνια, ιδιαίτερα στις πολυμερείς συζητήσεις και διαπραγματεύσεις, όπως το G20, όπως συζητήσεις για την κλιματική αλλαγή, όπως για τις άλλες διεθνείς ε, συζητήσεις και διαπραγματεύσεις, βήμα το βήμα μπορούμε να αναπτύξουμε μια κοινή θέση και μπορεί η Επιτροπή από πλευράς της να βοηθήσει έτσι ώστε να εκφραζόμαστε με μία φωνή, όπως ήδη το πράττουμε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Αυτό ήταν ε, όσο αφορούσε το δεύτερο κομμάτι της ερώτησης σας. Για το πρώτο. Η συνθήκη της Λισαβόνας έχει περιορίσει στην οριστική τους πλέον, ε, στον οριστικό τους αριθμό, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πλέον έχει κλείσει, έχει κλειδώσει ο αριθμός, δεν μπορεί να αλλάξει. Καθώς όμως δεν ε, κυρώθηκε εγκαίρως η συνθήκη της Λισαβόνας, οι εκλογές έγιναν με βάση την Ίκαια. Και έτσι στην ε, διάρκεια της θητείας θα ενταχθούν ακόμη 18 νέοι ευρωβουλευτές Οπότε πρέπει και να προσαρμοστούμε αναλόγως στις αλλαγές αυτές. Όμως από την επόμενη θητεία πάμε στους 715 σήμερα. Επίσης, όπως τα γνωρίζετε, υπάρχει συμφωνία από την τρέχουσα θητεία να αρχίσει να εφαρμόζεται νέο καθεστώς για τους ευρωβουλευτές, για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως επίσης και καθεστώς για τους βοηθούς των Ευρωβουλευτών. Το νέο αυτό καθεστώς, αντίθετα με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, πλέον χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Αυτό λοιπόν που πριν περνούσε από τον εθνικό κορβανά, τώρα χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό επίπεδο. Κύριος Σταφ. Με έκπληξη βλέπω ότι υπάρχει ενδεχόμενο να ενοχληθεί ο τύπος από την ενίσχυση του ρόλου αλλά και του επίπεδου εξυπηρέτησης και της ποιότητας ε, των ε, πραγματογνωμών των ειδικών που θα απασχολεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί τώρα με όλες τις νέες εξουσίες που έχουμε και την εκπροσώπησή μας σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα προφανώς και θα πρέπει να αναπτύξουμε δραστηριότητες και να έχουμε τους απαραίτητους ανθρώπινους πόρους και για τομεί στους οποίους μέχρι τώρα δεν είχαμε εξουσίε και δραστηριότητες. Όπως είναι η δικαιοσύνη. Τα εσωτερικά. Η εξωτερική πολιτική και η πολιτική άμυνα. Εάν λοιπόν δεν μπορούσαμε να επιδείξουμε ε, αποτελεσματικότητα, επαγγελματισμό θα έλεγα στους τομείς αυτούς, πρώτος ο τύπος θα μας ε, ε, επίπλητε. Επίση, θέλω να σημειώσω ότι στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων ήδη έχει εκτεταμένε του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχει συνεργασία εκτεταμένη με τι κοινέ επιτροπέ, παραδείγματι ε, της, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και των αντίστοιχων ε, επιτροπών μάλλον των Εθνικών Κοινοβουλίων των 27 κρατών μελών. Έχουμε τακτικέ επαφέ με ενδιαφέρουσε ανταλλαγέ απόψεων μεταξύ εκείνων και ημών. Επίσης, ε, θέματα χρηματοδότησης, στα οποία αναφέρθηκα και νωρίτερα. που θα αφορούν τομείς ασφάλειας και εξωτερικής, ε, άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, θα μπορέσουμε να τα φέρουμε σε διάλογο στις επαφές μας με τα Εθνικά Κοινοβούλια, που θα μπορούν και εκείνα να μιλήσουν. Παρακαλώ. Από τη Ραδιο Εσπανιόλα. Θα ήθελα να ρωτήσω συγκεκριμένα για τους 18 νέους ευρωβουλευτές. Ποια είναι η κατάσταση. Κάποια κράτη ήδη του έχουν επιλέξει, κάποια όχι. Πρέπει να έρθουν όλοι ταυτόχρονα, υπό ποιου όρου, από πότε αρχίζουν να, φτάνουν, να καταφτάνουν μάλλον στο κοινοβούλιο. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη συμφωνία. Δεχάν. μέχρι ότου ε, φτάσουμε να έχουμε θέμα ε, για συζήτηση στο Κοινοβούλιο, για έγκριση στο Κοινοβούλιο ε, για κείμενο επίπεδου συνθήκης, φερειπίν συνθήκη για την ένταξη Κροατίας, μέχρι τότε μπορούν να είναι παρατηρητές. Αυτή είναι η πρακτική που ακολουθήσαμε και στο παρελθόν με τα κράτη που ήταν υποψήφια και τα οποία μέχρι την ε, πλήρη τους ένταξη απέστελναν παρατηρητές εδώ στο Κοινοβούλιο. Τώρα, μέχρι ότου γίνουν πλήρη μέλη αυτά, αυτοί οι 18 νέοι ευρωβουλευτέ, νέα μέλη του Κοινοβουλίου, ασφαλώ από κάπου πρέπει να αντλήσουν την νομιμοποίησή του με κάποια μορφή εκλογική διαδικασία. Το πιο απλό και κάποια κράτη το διαθέτησαν ε, με νόμο, κάποια άλλα ίσως να βρουν διαφορετικό τρόπο, είναι να έλθει ο πρώτος στη λίστα, ο πρώτος επιλαχών από την αντίστοιχη μέχρι τώρα, από την τελευταία εκλογική λίστα. Όπου υπάρχει εθνική λίστα για ολόκληρη τη χώρα πρόβλημα δεν υπάρχει. Απλώς προσθέτουμε μία ακόμη δύο έδρες από εκείνους που δεν είχαν έρθει μέχρι τώρα. Από τα κράτη όμως που έχουν εκλογικές περιφέρειες, εξ όσων εγώ αντελήφθην πάλι για τα περισσότερα κράτη δεν υπάρχουν δυσκολίες, διότι η κατανομή των εδρών αναεκλογική περιφέρεια γίνεται επί της αναλογίας επί του πληθυσμού και άρα μπορούμε να πούμε σε βάση πληθυσμού ε, ποια ποσοστά ορίζουν την εκλογική περιφέρεια από την οποία θα έρθει ο εν λόγω ε, Υποψήφιο ευρωβουλευτής, δηλαδή Ποιο θα είχε εκλεγεί εάν υπήρχε μια, μια έδρα παραπάνω. Και ένα παράδειγμα μπορώ να σας δώσω από τη Γαλλία, για την οποία από ό,τι ξέρω δεν έχουν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα. Βλέπω, νομοθετικά δηλαδή, βλέπω ότι μάλλον προς αυτή τη λύση προσανατολίζεται. Παρά το γεγονό ότι ο εμπειρογνώμων επί του θέματος είναι ο Άντριου Νταφ, και επειδή και στην Επιτροπή μας θα πρέπει να συζητηθεί ένα ανάλογο ζήτημα, να σας πω εδώ ότι υπάρχουν τρία βασικά προβλήματα. Πρώτον, τα κράτη-μέλη πρέπει να κυρώσουν μέσω πρωτοκόλου και αυτό δεν θα διαρκέσει παραπάνω από ένα χρόνο, την εφαρμογή της συνθήκης της ε, Λισαβόνας για τους νέους αυτούς ευρωβουλευτές. Επομένως, οι 18 αυτοί ευρωβουλευτές θα μπορέσουν να ε, ενταχθούν όταν θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της ε, κύρωσης μέσω πρωτοκόλλου από όλα τα κράτη-μέλη. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να διαρκέσει μήνες, παρά το γεγονός ότι η Ισπανική Προεδρία έχει πρόθεση να χρησιμοποιήσετε μια διαδικασία που θα είναι το δυνατόν συντομότερο για το πρώτο εξάμεινο του 2010 αλλά επιμένω θα μπορούσε να διαρκέσει και για όλο το 2010. Το δεύτερο στοιχείο είναι πώς θα επιλέξουμε αυτά τα νέα πρόσωπα. Η πλειονότητα των χωρών, όπως είπε ο Ζανλουκ Λουκ είναι χώρες οι οποίες έχουν ήδη καθορίσει ποιοι θα είναι οι επιπλέον υποψήφοι. Ε, αλλά το πρόβλημα είναι ότι κάποιες χώρες έχουν ένα νομικό σύστημα ε, πιστοποίησης αν θέλετε των εδρών, αλλά κάποιες ε, χώρες όχι. Ε, στη Γαλλία για παράδειγμα δεν έχει ρυθμιστεί ακόμα το ζήτημα, αλλά την περασμένη εβδομάδα στην Ολομέλεια του Στρασβούργου πέρασε ένα πολύ σημαντικό θέμα, στο οποίο καθοριζόταν το πώ θα εντοχθούν οι νέοι ευρωβουλευτέ. και εκεί είχαμε μια τροπολογία την οποία παρουσίασε ο κύριος Ντόαφ εξ ονόματος των φιλελευθέρων και εμείς ε, ε ως και στην τροπολογία αυτή ζητούσαμε οι νέοι ευρωβουλευτέ οι οποίοι αντιστοιχούν σε 18 άτομα να προέρχονται ούτως ή άλλως ε, από τις ε, ε, από τους καταλόγους, από τις λίστες ε, των ευρωεκλογών του Ιουνίου και αυτή η τροπολογία απορρίφθηκε. Ε, υπήρχε μια λογική ε, προερχόμενη από τη Γαλλία, όπως είπε ο κ. Ντεάν, που έλεγε ότι το δικό τους σύστημα δεν τους επιτρέπεται να τους επιλέξει μέσω των εκλογικών καταλόγων, μέσω της λίστας που είχαν σε ευρωεκλογές και θέλουν ένα σύστημα το οποίο θα είναι πιο ακριβές για να επιλέξουν τους ε, επιπλέον ε, ε, βουλευτές. Νομίζω ότι η Γαλλία έχει ένα ή δύο νέους βουλευτές. Έχει λοιπόν άλλους δύο. Και τελικά πέρασε αυτή η θέση, διότι τη στήριξε το ΕΛΚ και γιατί ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον οποίο εγκρίναμε την περασμένη Πέμπτη, δεν καθορίζει ότι η διαδικασία εκλογές θα πρέπει να είναι πανομοιότυπος και να καθορίζεται από τις λίστες του Ιουνίου. Και έχουμε και το τρίτο πρόβλημα, το πρόβλημα των παρατηρητών, που είναι αν θέλετε η ενδιάμεση φιγούρα. Μόνο το κοινοβούλιο θα μπορέσει να αποφασίσει πότε και πώς θα πρέπει να ενσωματωθούν. Ε, φυσικά υπάρχει περίπτωση να σωματοθούν μουτάντι μουτάντι, όπως λέει το άρθρο, με την ίδια διαδικασία με την οποία ακολουθήθηκε για άλλες χώρες ε, οι οποίες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι να έχουμε την πλήρη ένταξη. Επομένω, θα πρέπει να δημιουργηθεί το καθεστώς παρατηρητή από το Προεδρείο του Κοινοβουλίου. Ε, αλλά υπάρχουν τρία διαδοχικά βήματα τα οποία πρέπει να ε, γίνουν όπως σας εξήγησα. Επόμενη ερώτηση. have political because uh, I'm just thinking this whole story. Θα ήθελα να ρωτήσω ε, για το θέμα των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί δεν ξέρω αν μπορώ να πείσω τους αναγνώστες μου θα είναι πιο κοινωνικό, πιο υπέρ της προστασίας του καταναλωτή, θα είναι πιο φιλικό προς επιχειρήσεις στο Κοινοβούλιο, θα ανοίξει περισσότερο τις πύλες του για τους μετανάστες, θα είναι πιο ανοιχτό προς μετανάστες ή το αντίθετο. Τι περιμένετε από τη στάση περιμένετε ότι θα κρατήσει το Κοινοβούλιο σε αυτούς τους τομείς. Ah, um, Κύριε Σταφ, η πιο απλή απάντηση που μπορώ να είναι ότι εξαρτάται αυτό από την ισορροπία των πολιτικών δυνάμεων μέσα στο Κοινοβούλιο. Προφανώς, αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι στη διαδικασία της συναπόφασης χρειάζεται συχνά να ληφθεί μια απόφαση με την ενισχυμένη, με την ειδική πλειοψηφία. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνήσουν οι βουλευτές ανεξαρτήτως των της πολιτικής ομάδας ή πρέπει να συμφωνήσουν περισσότερες πολιτικές ομάδες για να ληφθεί μια απόφαση. Και αυτό σας το λέω ως κάποιος από την ομάδα των φιλελευθέρων που βρίσκεται στο κέντρο ουσιαστικά, βρίσκεται ακριβώς στα μισά του Κοινοβουλίου. θέματα εργασιακά επί παραδείγματι πολλές φορές έχουν ε, υποστηριχθεί από κάθε πτέρυγα του Κοινοβουλίου προς τη μία κατεύθυνση, ενώ σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να ακολουθηθεί μια διαφορετική τάση. Υπάρχουν τομείς από τους οποίους ακόμη δεν έχουμε εμπειρία. Και το να αναλάβουμε παραδείγματα για τη γεωργική πολιτική για πρώτη φορά εξουσίες λήψη αποφάσεων, ασφαλώς θα επηρεάσει σημαντικά το χαρακτήρα της Επιτροπής Γεωργίας και δεν θα είναι πλέον μια επιτροπή στην οποία εδρεύουν μόνο ε, γεωργοί και κτηνοτρόφοι, τους οποίους κατά τα άλλα βρίσκω αλλά δεν θα είναι μόνο αυτοί οι μέλη της Επιτροπής Γεωργίας. Όπως επίσης, φαντάζομαι, πως η Επιτροπή Πολιτισμού, η Επιτροπή Γεωργίας θα ε, προσελκύσει ως μέλη και κάποιους έξω από τη Γεωργία, τον επαγγελματικό χώρο της Γεωργίας, που θέλουν να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων για τα Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η αλλαγή θα επισύμβει από τη μία μέρα στην άλλη, θα δούμε, πιστεύω, ποιοτική βελτίωση τις στάσεις του Κοινοβουλίου ε, στους τομείς όπου ενισχύονται οι εξουσίες μας. Ήταν πολύ εύστοχη η ερώτησή σας. Την απάντηση θα μας τη δώσει ο χρόνος. Νομίζω ότι έχουμε περιθώριο για μια ακόμη δύο ερωτήσεις. Πριν με αφήσουν κατά μόναχο οι συνάδελφοι εδώ πάνω στο Προεδρείο. Παρακαλώ. Από το Χρούν Άμστερνταμ, ε, ε, ε, το περιοδικό από τις χώρες στην Ολλανδία. Θα ήθελα να ρωτήσω για την συνθήκη της Λισαβόνας. Θεωρείτε ότι μπορεί να αποτελέσει αναγνώριση από πλευράς του Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου ως νομοθετικού σώματος, ενώ ταυτόχρονα το Συμβούλιο μάλλον σπέβδει να λαμβάνει αποφάσεις ε, για το SWIFT, για το πρόγραμμα Στοκχόλμης και κλεισμένο των θυρών χωρίς σύμπραξη του Κοινοβουλίου. Πώς δηλαδή κρίνεται την προσέγγιση αυτού του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πώς διαβλέπετε την εξέλιξη των σχέσεων στο μέλλον. Είναι σαφές ότι η συνθήκη της Λισαβόνας και για πρώτη φορά στο ίδιο το κείμενο της συνθήκης ο ορισμός ε, των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου και εδώ μιλάω για το Συμβούλιο και όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Οι αρμοδιότητες λοιπόν του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου καθορίζονται με ακριβώς τους ίδιους όρους. Για πρώτη φορά λοιπόν η συνθήκη παρουσιάζει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σαν τις δύο βουλές, αν θέλετε, που έχουν νομοθετικό έργο. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να γίνουν προσαρμογές στο Κοινοβούλιο, αλλά ακόμα πιο σαφές είναι το γεγονός ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να εργάζεται πλέον με διαφορετικό τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, Στην έκθεσή μου, στην οποία αναφέρθηκε και ο Άντριου, επεσήμανα την ανάγκη να υπάρχει ένα πραγματικό Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, το οποίο θα είναι διαφορετικό από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Τώρα πολύ συχνά γίνονται την ίδια μέρα με τους ίδιους ανθρώπους και στην ίδια συνεδρίαση τα θέματα αυτά. ο συντονισμός του έργου του Συμβουλίου με το Κοινοβούλιο θα πρέπει να, θα είναι μάλλον η νέα πρόκληση ε, που προκύπτει από τη συνθήκη. Και αν το Συμβούλιο δεν οργανωθεί ώστε να το επιτύχει, τότε αυτό σε πρώτη φάση τουλάχιστον θα είναι δύσκολο. Ε, και είμαι βέβαιος ότι και αυτοί θα μάθουν από τη διαδικασία και διαπιστώνω ότι πρέπει να μάθουν και να εντάξουν κάποια νέα στοιχεία. Επί να σας πω κάποια πράγματα εσωτερικά αν θέλετε, κάποια, μια μέρα να σημειώνω κάποια πράγματα για την ε, υπηρεσία εξωτερικών θεμάτων. Μιλούν πάτε για τον είπα το εκπρόσωπο και ξεχνούν ότι είναι αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει να το μάθουν αυτό. Έχει δίκαιο, λέει ο κύριος Τάφ. Μια τελευταία ερώτηση, παρακαλώ. Είμαι από την Ελλάδα, από το νησί Ζάκυνθος και θέλω να ρωτήσω ε, πώς η νέα Ευρώπη θα επηρεάσει τις αποφάσεις της νομοθετικά όσον αφορά τα τροποποιημένα τρόφιμα και γενικά τους μεταλλαγμένους χαρακτήρες των τροφίμων τα οποία κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά. Θα υπάρχει κοινή νομοθετική γραμμή ή κάθε χώρα θα λαμβάνει υπόψη της τα δεδομένα τα βιομηχανικά και τα εμπορικά για να αφήσει όπως αυτή τη στιγμή ανεξέλεκτα μεταλλαγμένα τρόφιμα να κυκλοφορούν. Um, the uh, position on uh, GMOs. Η γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί και η θέση μας από αυτού επαναξιολογούνται αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα υπάρξει μια νέα πρόταση την Άνοιξη. Και θα πρέπει να περιμένουμε λοιπόν να δούμε ποια είναι η πρόταση και από εκεί και πέρα το Κοινοβούλιο θα πρέπει να καθορίσει και τη θέση του ε, σε εκείνη τη φάση. Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη γιατί πρέπει να φύγω και εγώ τώρα. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ και απολαύστε τη νέα συνθήκη. Thank uh, We will do now a break. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα τώρα, πέντε λεπτάκια και θα ξεκινήσουμε με το δεύτερο τμήμα του σεμιναρίου. Ευχαριστώ, Άντριου. Εκεί ο Σοβανός, ας πούμε, ο Δανιάς, ο οποίος επιλέγει. Μέσα από το